ανταποκριθεί επιτέλους στις απαιτήσει του Κοινοβουλίου. Χρειάζεται μια εντατική συζήτηση και έχει φτάσει η ώρα να γίνει αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω λάβει από τον ε, κύριο Λουίτζι Ντε τη αίτηση προάσπιση τη ασυλία του και των προνομίων του στο πλαίσιο δικαστική δίωξη που εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου του Καταντζάρο. Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφο 3 του κανονισμού, η αίτηση παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή νομικών θεμάτων. Έχω λάβει από το Συμβούλιο επίση άλλη ανακοίνωση αυτή. Ε, τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση μαζί με το σκεπτικό που το οδήγησε στην έγκρισή τη, καθώ και την θέση τη επιτροπή. Ο τίτλο θα ανακοινωθεί στα πρακτικά τη παρούσα συνεδρίαση. Η προθεσμία των τριών μηνών, την οποία διαθέτει το Κοινοβούλιο προκειμένου να αποφανθεί, αρχίζει αρχίζει από αύριο, 25 Μαρτίου 2011. Τα συνοπτικά πρακτικά αυτή και τη θεσινή συνεδρίαση θα υποβληθούν προ έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή τη επόμενη περίοδου Συνόδου αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα διαβιβάσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση στα πρόσωπα και του φορεί που αναφέρονται σε αυτά. Διακόπτεται η Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση λίγη. Καλό μεσημέρι σε όλους.